ερώτηση προ την Επιτροπή όσον αφορά την θαλιδομίδη. Πρώτα απ' όλα, Κονζάλες Πόνς. Εκτός μικροφώνου αρχίζω, μιλητής. Γιατί, γιατί είναι θελιδομίδη, γιατί είναι ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί και χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια μέχρι το 1961, γιατί δημιουργεί ε, κακή διαμόρφωση του εμβρίου και γιατί κανείς δεν ε, φρόντισε να μην κυκλοφορήσει μεταξύ των εγγύων γυναικών. Πολλοί γυναικολόγοι, βέβαια, επειδή συνταγογραφούσαν το φάρμακο αυτό, έπαιρναν δώρα. Πάνω από 10.000 παιδιά, χωρίς χέρια ή πόδια ή με μικρότερα από το κανονικό γεννήθηκαν. Και φαίνεται σαν να είναι ψέμα, αλλά είναι αλήθεια. Τα θύματα χρειάστηκε να περιμένουν 50 χρόνια μέχρι να του ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Γιατί οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών έκλειναν τα μάτια. Γιατί είναι η μεγαλύτερη υγειονομική τραγωδία στην ευρωπαϊκή ιστορία. Γιατί οι μητέρε που πήραν το φάρμακο αυτό, που το, το συντογράφησαν οι γιατροί του, ένιωσαν ενοχέ και πολλέ, ακόμα, σε πολύ μεγάλη ηλικία βέβαια, εξακολουθούν να νιώθουν τι ενοχές αυτέ, χωρί κανεί να γυρίσει και να του πει δεν φταίτε οι μανάδες αυτές είναι αθώες και κανείς δεν αγαπάει περισσότερο τα παιδιά τους από ότι αυτές οι ίδιες. Ποτέ δεν έγινε τέτοια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα. Είμαστε μπροστά σε ένα ανθρώπινο δράμα το οποίο απαιτεί μια πολιτική λύση γιατί μας κάνει να τρεπόμαστε 50 χρόνια μετά να μην έχει υπάρξει πολιτική λύση. Γιατί στη χώρα μου υπό το Φράκο και τη δικτατορία το φάρμακο αυτό αποσύρθηκε με καθυστέρηση τριών ετών γιατί στην Ισπανία είχαμε 500 θύματα και μόνο 24 αναγνωρίστηκαν. Γιατί στην Ισπανία καμία κυβέρνηση, κανένα κόμματο, ούτε οι κυβερνήσει του δικού κόμματο δεν θέλησαν να λύσουν τα προβλήματα αυτά όλων εκείνων που ήταν θύματα του φαρμάκου αυτού γιατί στην Ισπανία τα θύματα τα έκρυψε η δικτατορία και τα ξέχασε η δημοκρατία. Γιατί τα βαντεμέκουμ περιλαμβάνουν φάρμακα με θαλιδομήν μέχρι το 1950. Γιατί όλοι από τη δικιά μου τη γενιά θα μπορούσαμε να είμαστε θύματα της θαλιδομίδης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να πιέσει και τη γερμανική κυβέρνηση και την ισπανική κυβέρνηση. Εγώ ποτέ δεν ένιωσα περισσότερο ασφαλής από τότε που άρχισα να υποστηρίζω τα θέματα από εδώ, από αυτή την έδρα. Τα θύματα πρέπει να έχουν κάποια βοήθεια. Μέχρι τώρα χειροτερεύει η κατάστασή τους χωρίς καμία επανόρθωση, καμία αποζημίωση. Σήμερα είναι βέβαια αργά για να διορθωθεί ο πόνος. Θα ήταν όμως δίκαιο να γίνει κάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ο μιλητής, ο κύριος Κρότε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πράγματι λυπηρό το ότι συζητάμε αυτό το πράγμα σήμερα τόσο καιρό μετά το σκάνδαλο της ε, Θαλιδομίδης ότι έχουμε 900 θύματα που δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί σωστά και δεν υπάρχει καμία λύση στο τέλος της ημέρας και ευχαριστώ τον Επιτροπό που βρίσκεται εδώ πέρα σήμερα μαζί μας για να ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις των κρατών μελών που επέτρεψαν να κυκλοφορήσει το φάρμακο και έδωσαν άδεια. Πρέπει να υπάρξει μια αποζημίωση και ο χρόνος πιέζει. Γιατί κάθε μέρα τα θύματα παλεύουν με την καθημερινότητα. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε πίεση να στείλουμε ένα μήνυμα στις πρωτεύουσε των κρατών που ε, αφορά το σκάνδαλο αυτό και όπου ζουν οι άνθρωποι. Και πρέπει να πω πως το να ρίχνει ο ένας ή ε, μία χώρα το φταίξιμο στην άλλη δεν ωφελεί σε τίποτα τα θύματα. Καλό είναι να στείλουμε ένα μήνυμα ενωμένοι ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή λύση για αυτούς οι οποίοι δεν αποζημιώθηκαν από το σχετικό ίδρυμα στην ε, Γερμανία. Και αναμένω πραγματικά την αντίδραση του Συμβουλίου. Δυστυχώς τα έδρανα του Συμβουλίου είναι άδεια. Εγώ θα ήθελα να είναι εκεί πέρα κάποια κράτη-μέλη για να ακούσουν αυτά που έχουμε να πούμε αλλά ίσως δεν ξέρω να στείλουμε το πρώτο μήνυμα και να μην χαλαρώσουμε, να συνεχίσουμε να παλεύουμε για τους 900 αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί επαρκώς. Για να αποζημιωθούν και να βρουν το δίκαιο τους σε τελική ανάλυση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλοί πιστεύουν ότι το θέμα της θαλιδομίδης είναι παρελθόν. Κάτι που συνέβη στα μέσα του 20ου αιώνα και τελείωσε. Φυσικά αυτό είναι εντελώς λάθος. Οι επιπτώσεις θαλιδομίδης δεν είναι απλώς ιστορικής σημασίας. Εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα και να τις βλέπουμε. Πολλοί επιζώντες και οι οικογένειές τους ε, σε όλη την Ευρώπη έζησαν άθλια ε, επί 50 χρόνια και ακόμα έχουν προβλήματα καθημερινά οικονομικά, δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος περίθαλψής τους, δεν θέλουν να ζήσουν μια πολυτελή ζωή. Θέλουν απλώς αρκετά ε, για να ζουν άνετα, να μην έχουν ανησυχίε και χρόνιους πόνους. Αυτοί που δουλεύουν ακόμα ε, δυσκολεύονται πράγμα πολύ να δουλεύουν 100%. Η κινητικότητά τους ε, επιδεινώνεται και συχνά πέρα από τα φυσικά προβλήματα που έχουν, τα προβλήματα τα σωματικά έχουν και κατάθλιψη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τη βοήθεια. Πολλέ χώρε στην Ευρώπη αντιμετώπισαν το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο. Στη Γερμανία η κυβέρνηση ε, δίνει λεφτά ε, μέσω του Ιδρύματο Κοντέργαν ε, στι οικογένειε. Και αυτό είναι μια αναγνώριση τη ευθύνη. Τι έχουν κάνει όμω όλοι οι υπόλοιποι στην Ευρώπη, τα υπόλοιπα θύματα που έχουν λάβει ελάχιστα χρήματα ή τίποτα. Περιμένουν ακόμα η γερμανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και να αναλάβει τι ευθύνε τη και να δώσει το, τα μικρά αυτά ποσά τα οποία όλο και μειώνονται από χρόνο σε χρόνο. Γιατί λοιπόν θέσαμε αυτό το πρόβλημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μένα είναι σαν να λέμε στην Κομισιόν. Κύριε Αντρικάητε, βοηθήστε μας, ούτε ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα για να υπάρξει μια συμφωνία και που θα αφορά όλους όλα τα θύματα, ούτως ώστε να ζήσουν τη ζωή τους με άνεση, ε, την οποία δεν είχαν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπεθέρα Μπαστερετσέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε πίτροπε, είναι εξωπρόσεχτο ότι σήμερα συζητάμε στην Ολομέλεια Πράγματα τα οποία έλαβαν χώρα πριν από περισσότερο από 50 χρόνια. Σήμερα τα θύματα εξακολουθούν να υποφέρουν από τις συνέπειες. Πολλοί πολίτες που μας ε, παρακολουθούν θα αναρωτιούνται «Μα τι έγινε τόσο όλο αυτό τον καιρό». Η απάντηση είναι ότι 50 χρόνια αργότερα πολλά από τα θύματα της ε, Θαλιδομίδης ζητούν δικαιοσύνη, ζητούν την εγγύηση να έχουν μια ζωή με αξιοπρέπεια. Η τραγωδία αυτή της Θαλιδομίδης άλυξε την ιστορία της Υπήρου μας. Επέτρεψε να εγκριθεί νομοθεσία η οποία μας επιτρέπει περισσότερη ασφάλεια από τα φάρμακα. Χάρη σε αυτό αποφεύγουμε νέες τέτοιες καταστροφές εξαιτία φαρμάκων. Όμως, δεν προχώρησε εξίσου και η επανόρθωση, η αποζημίωση όλων αυτών των θυμάτων, παιδιών. Παρ' όλα αυτά κοστέζουν πολύ η βοήθεια, η θεραπεία και πολλοί πολίτες δεν καταφέρνουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Το 1972 δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Κοντεργάν που μετά από ένα νόμο που εκαθιδρεί την οικουμενικότητα των βοηθειών. Όμως στη Γερμανία έχουν αναγνωριστεί 3.000 θύματα, στην Ισπανία ένα μόνο. Σε άλλε χώρες έχουν γίνει πολλά από τις κυβερνήσει, ακόμα και στην Αυστραλία. Ενώ στην ε, Ισπανία κανεί δεν θυμάται τα θύματα αυτά. Τους έχουν εγκαταλείψει στην τύχη τους και έχουν περιθεριοποιεί. Κατά τη δικιά μου την κοινοβουλευτική δραστηριότητα γνώρισα από πρώτο χέρι την ιστορία αυτών των ανθρώπων και μίλησα με μέλη τη ΑΒΙΤΕ που είναι η Ισπανική Οργάνωση Θυμάτων Θαλιδομήνη πρέπει να αναγνωριστούν τα θύματα. Ήρθε η ώρα να υπάρξει μια συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακριβώς ζητά και η προφορική μας ερώτηση, βάσει της οποίας όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν υποστεί την θαλιδομίδη και τα αποτελέσματά της πρέπει να αποζημιωθούν. Δεν θέλουμε άλλη καθυστέρηση. Είναι δίκαιο να γίνει κάτι τέτοιο και δεν είναι σωστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο Εκ. κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, βεβαίω ε, το θέμα αυτό είναι η πιο γνωστή καταστροφή της φαρμακευτικής ε, βιομηχανίας. Αφού δοκιμάστηκε σε ζώα, βλέπουμε και πάλι γενικώ πειράματα σε ζώα. Και μετά τα αρχικά πειράματα, η γερμανική εταιρεία Contagan το βγάλε αυτό στην αγορά ως προϊόν ασφαλές ε, για έγκυες και ε, έμβρια παρά το ότι βεβαίως δεν είχαν γίνει πειράματα σχετικά. Μιλάμε για παγκοσμίω 5 με 10.000 άτομα που γεννήθηκαν με δυσπλασίες ε, συγγενείς. Έχουν λοιπόν αποζημιωθεί κάποια άτομα, κάποια άλλα όχι, δεν έχουν καν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να αναλάβει το ηθικό βάρος, να βοηθήσει όλους ε, τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, να τους ε, αποζημιώσει και να έχουν βεβαίως πρόσβαση σε ε, βοήθεια στο σπίτι. Έχουν επίσης δικαίωμα στο να ζουν ανεμπόδιστα. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος πως η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μια κοινή αγορά για τις φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να έχει και ένα κοινό σύστημα για καταστροφές φαρμακευτικές. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι σήμερα αρμοδιότητα της Ένωσης. Επίσης, ως μέλος της Επιτροπής ΕΝΒΗ πρέπει η Κομισιόν, θεωρώ, και το Συμβούλιο να ζητήσουν αυστηρότερη τήρηση των κανόνων και μεγαλύτερη ευθύνη για τις εταιρείες οι οποίες φέρνουν τα προϊόντα αυτά στην αγορά. Χρειάζεται βεβαίω και κοινωνική αποδοχή, αλλά πάνω απ' όλα δικαιοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσουμε γι' αυτό. Κύριε Αντριουκάητης, ο Βίλι Μπραντ, ο πρώην καγκελάριος, είχε πει πως η πολιτική χρειάζεται μια ηθική βάση. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Evans. Κύριος Η κυρία Evans. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί πολλά χρόνια οι επιζώντες της Θαλιδομίδης ζήτησαν δικαιοσύνη. Αυτοί που είναι στη δική μου εκλογική περιφέρεια και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς έχουν όλο και περισσότερες ανάγκες ε, υγείας, ε, υψώνουν τη φωνή τους και εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να αναλάβουμε δράση η οποία έχει καθυστερήσει. Ξέρουμε ότι η εκστρατεία συνεχίζεται, ούτως ώστε να χυθεί άπλετο φως για το ρόλο της γερμανικής κυβέρνησης στην ε, πρόορη, ε, στο πρό, ε, πρώιμο τέλος της δίκης ε, της δεκαετίας του 1970. Τελείωσε γρήγορα η δίκη και έκρυψαν διάφορα αποδεικτικά στοιχεία και έτσι δεν μπορούσαν να ζητήσουν ε, τα, τις αποζημιώσεις στα θύματα για να καλύψουν ε, τα προβλήματα διαβίου. Κάποιοι επιζώντες έλαβαν κάποια οικονομική στήριξη, αλλά άλλοι τίποτα. Θέλουμε δικαιοσύνη και ισότητα για όλους τους επιζώντες σε όλες τις χώρες. Όπως ως αιρετή εκπροσωπή τους θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι και οι σημερινές και οι μελλοντικές ανάγκες τους καλύπτονται. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να το εξασφαλίσει αυτό. Ήδη περίμεναν πάνω από 50 χρόνια. Πιστεύαμε, πιστεύουμε ότι 10.000 παιδιά τουλάχιστον σε όλο τον κόσμο έχουν επηρεαστεί από την θαλίδομίδη. Αλλά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο. Επίσης ε, υπάρχουν στοιχεία για τις αυξημένες ανάγκες υγείας, για την οδύνη, τον πόνο. Ε, έχουν γίνει μελέτες στο, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο που δείχνει πόσο επιτακτικές είναι οι ανάγκες αυτές. Επίσης, επίσης υπήρχε διαπαραταξιακή στήριξη εδώ στο Κοινοβούλιο για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτό τον αγώνα που κράτησε πάνω από 50 χρόνια. Νομίζω ότι είναι και η ώρα για να αποδώσουμε δικαιοσύνη ε, σε κάτι το οποίο ψοβεί σε ένα πρόβλημα το οποίο σοβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κυρία Τζέιμς, θέλω να χαιρετήσω όλα τα θύματα της Αλιδομίδης σε όλη την Ευρώπη για την επίμονη ε, προσήλωσή του στην εκστρατεία αυτή. Το, Μάιο του 2015, πριν από 9 μήνες, όλοι οι ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα και τα, τις ομάδες επέμειναν ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο σκάνδαλο ε, για την ε, απόλυτη αδράνεια που υπάρχει. Ε, είναι σχεδόν ε, το πρόβλημα 60 ετών. Επί 60 χρόνια η γερμανική κυβέρνηση και η εν λόγω φαρμακευτική εταιρεία έκαναν ό,τι μπορούσαν, καθυστέρησαν, ε, κέρδισαν χρόνο ούτως ώστε να αποφύγουν να καλύψουν τις ανάγκες των θυμάτων. Όλες οι οργανώσεις ε, ντρέπονται για τις δράσεις τους κατέφυγαν σε κάθε δικαιολογία, παραθυράκι, χρησιμοποίησαν όλες τις τακτικές ε, καθυστερήσεις για να αποφύγουν να δοθεί ε, μία λύση και να δοθεί αποζημίωση. Είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Τα θύματα, ορισμένοι από αυτούς είναι πάρα πολύ ανάπηρα, παρόλα αυτά είναι άνθρωποι και αυτά και θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Ζητούν ε, ένα επαρκές και εύλογο ποσό, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά του. Ε, και μάλιστα καθώ γυράσκουν είναι και περισσότερα τα προβλήματα και δεν θα πρέπει να του αγνοήσουμε. Για ένα, για ένα θεσμικό όργανο το οποίο ε, υπερασπίζεται του, τις μισθολογικές απαιτήσεις ε, των μη αναπήρων, γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρούμε ένα Υπάρχει και χρηματικό ποσό που θα επιτρέψει και στα θύματα της Θαλιδομίδης να ζήσουν τη ζωή τους όσο μπορούν πιο αξιοπρεπώς, όσο του επιτρέπει η αναπηρία. Απαιτώ από το Συμβούλιο, την Κομισιόν και τους Ευρωβουλευτές να επιβάλλουν κυρώσεις στην γερμανική κυβέρνηση για αυτή την απάνθρωπη, ε, σκληρή και περιπτή καθυστέρηση. Εννιά μήνες είναι πολύ ε, μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά 60 χρόνια είναι απαράδεκτο. Ο Επίτροπος Αντριουκάητης έχει το λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω εδώ σήμερα. Η καταστροφή της μας υπενθυμίζει σήμερα και πάντα θα μας υπενθυμίζει τις πιθανώς τραγικές συνέπειες που έχει η έλλειψη του ορθού ρυθμιστικού πλαισίου για τα φάρμακα. Η καταστροφή αυτή όμως κατέληξε στην φαρμακευτική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από 50 χρόνια σε μια συμφωνία για εναρμονισμένους ελέγχους και ένα υψηλό επίπεδο προστασία τη δημοσίευση. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε πριν από 60 χρόνια. Υπάρχουν όμω πάρα πολλοί επιζώντες που υφίστανται τι συνέπειε. Επιζώντες οι οποίοι χρειάζονται ηθική, κοινωνική και οικονομική στήριξη καθώς η ιατρική τους κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Πολλοί ευρωβουλευτές μου απίφθηναν επιστολή σε μένα προσωπικά και στην Επιτροπή τονίζοντας το θέμα. Έχω συναντήσει θύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Σουηδία πέρσι στις Βρυξέλλες και συζήτησα μαζί τους τα αιτήματά τους. Αναγνωρίζει την ανάγκη να βρεθεί μια κατάλληλη λύση για όλους τους επιζώντες που θα διασφαλίζει μια ποιότητα ζωής. Και έχω αναλάβει διάφορα, διάφορες σχετικές πρωτοβουλίες. Το Σεπτέμβριο του 2015 ενημέρωσα τις κυβερνήσεις πέντε χωρών για τις ε, συναντήσεις μου αυτές με στόχο να τις ενημερώσω. Θα ήθελα και πάλι να τους ευχαριστήσω που δέχτηκαν την πρόσκλησή μου να έρθουν σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια της φαρμακευτικής νομοθεσίας και βεβαίως ε, να μιλήσουν σχετικά. Επίσης, ε, τους ε, κάλεσα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε το ζήτημα. Επίσης, συζήτησα αυτό το θέμα πολλές φορές από όταν ξεκίνησε η θητεία μου με ενώσεις φαρμακευτικών εταιριών. Πριν από λίγες εβδομάδες μίλησα και στο Κοινοβούλιο για τις κλινικές δοκίμες όπως ξέρετε, θέμα που σχετίζεται με το σημερινό μας θέμα και θα ήθελα οι φαρμακευτικές βιομηχανίες να αναλάβουν περισσότερο τις ευθύνες τους. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης, οι οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών υγείας ε, και η διαχείριση των σχετικών πόρων είναι υπόθεση των κρατών μελών. Όπως όλοι γνωρίζουμε και οι αποζημιώσεις αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Οπότε η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να συστήσει ένα πλαίσιο αποζημίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί μόνο να εκφράσει την υποστήριξή της για την εξέβρεση πολιτικής λύσης στο εθνικό επίπεδο μέσω της συνεργασίας. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω εσάς, τους βουλευτές, να μεταφέρετε στις εθνικές σας κυβερνήσεις τις ειδικέ ανάγκες των θυμάτων της Θαλιδομίδης και την ανάγκη να στηριχθεί το θέμα αυτό. Τέλος, να υπογραμμίσω ξανά την κοινωνική ευθύνη της φαρμακοβιομηχανίας να στηρίξει τα θύματα. όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις. Ευχαριστώ, κύριε Επιτροπέ. Και τώρα, από το Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Μικολάσιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 60 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόκειται για ένα φάρμακο το οποίο ξεκίνησε να πωλείται πριν από 60 χρόνια με την εμπορική ονομασία Κονταγκάν όχι μόνο στην Γερμανία αλλά σε πάνω από 50 χώρες ε, παγκοσμίω ε, και σε πολλές ευρωπαϊκές και υπήρχαν βεβαίως ε, οι γνωστές παρενέργειες. Γνωρίζουμε πως ήταν φοβερές οι συνέπειες στα έμβρια δυσπλασίες ε, στα άκρα κυρίως αλλά και τα εσωτερικά όργανα, η καρδιά, όλα επηρεάστηκαν από αυτό το φάρμακο το οποίο το χρησιμοποιούσαν για να καταπολεμήσουν τους πονοκεφάλους ή την πρωινή ναυτία των εγγύων. Λοιπόν, Λυπούμε για το ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποιος ε, τρόπος για να αποζημιωθούν τα θύματα. Όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά χιλιάδες ε, είναι τα θύματα παγκοσμίως. Και όπως είπαμε πολλά ήταν τα θύματα αυτού του φαρμάκου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Καμπεθόν Ρουίθ. Η κυρία Καμπεθόν Ρουίθ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κρίση της θελιδομίδης ήταν τόσο σοβαρή που οδήγησε στο να αλλάξουμε την, φαρκο, την φαρμακοεπαγρύπνηση στην Ευρώπη. Αλλά 500 στην Ισπανία, άλλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Σουηδία δεν αποζημιώθηκαν ποτέ, εξακολουθούν να υποφέρουν και νιώθουν ότι τους έχουμε ξεχάσει πρέπει να παρακολουθήσουμε και να αποδώσουμε ευθύνες και στην φαρμακευτική εταιρεία, αλλά και ηθικά οι χώρε μέλη πρέπει να βοηθήσουν τα θύματα. Και αυτό ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συντονίσει την απάντηση αυτή που πρέπει να δοθεί στα θύματα. Στην Ισπανία το 2010 η σοσιαλιστική κυβέρνηση με ένα διάταγμα αναγνώρισε τα θύματα και προσπάθησε να τους δώσει μια κάποια αποζημίωση. Αλλά Μέχρι σήμερα φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετό αυτό. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω και κάνω έκκληση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να υπάρξει συντονισμό μεταξύ των χωρών μελών και από την Ευρώπη με τι χώρε μέλη να δώσουμε μια απάντηση δίκαια, σωστή και κατάλληλη στα θύματα αυτά. Εκ μέρου των Πρασίνων, η κυρία Ριβαζή έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είπατε ότι είναι ευθύνη των χωρών μελών να αποζημιώνουν τα θύματα. Όμως δεν μιλάτε για μια οδηγία που έχει να κάνει με το θέμα. Ούτε οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτή μου κάνει εντύπωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ελαττωματικά προϊόντα το 1985. Πρέπει να αναφερθεί η οδηγία αυτή. Γιατί? Γιατί αναφέρεται σε προθεσμίες που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα πια το θύμα μπορεί να δράσει μέσα σε τρία χρόνια από τότε που έλαβε γνώση της βλάβης που υπέστη. Και αυτό δέκα χρόνια το πολύ από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το φάρμακο. Μα οι προθεσμίες αυτές είναι πάρα πολύ μικρές. Και σε τι οδηγούν. Αναφερθήκαμε στην Ισπανία. Είναι τραγικό το σκάνδαλο αυτό της ε, θαλιδομίδης. 180 θύματα πήγαν στα νότατα δικαστήρια αλλά εξαιτία τη οδηγία αυτή του 85, τα δικαστήρια έκριναν ότι έχει παραγραφεί το αδίκημα. Και άρα τα θύματα δεν μπόρεσαν να πάρουν καμία αποζημίωση ούτε από το Κρούνανταλ, εργατεστήριο αυτό δηλαδή, το οποίο παρήγαγε την θελιδομίδη. Δεν είναι θέμα λοιπόν αυτό χωρών μελών, είναι πρόβλημα με την οδηγία που ψηφίσαμε εμεί το 85. Δεύτερον, στην οδηγία αυτή του 85 λέει ότι τα θύματα πρέπει να αποδεικνύουν ότι υπάρχει σχέση αίτιου και αιτιατού ανάμεσα στο φάρμακο και την ασθένειά τους. Μετά από το σκάνδαλο όμως αυτό της θελιδομίδης, τι έκαναν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί έκαναν την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Ε, αυτό πρέπει να κάνουμε και εδώ με την οδηγία μας αυτή όταν την αναθεωρήσουμε. Και τρίτον, άπαξ και ένα θύμα. Έχει ένα επίπτωση από το φάρμακο παρενέργειες από το φάρμακο. Εσείς ε, ξέρετε από τέτοια εργαστήρια πρέπει να τα πιέσουμε ώστε να αποζημιώνουν και στην περίπτωση αυτή παρενεργειών. Και αυτό είναι αρμοδιότητα της Ευρώπης κύριε Επίτροπε. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Από το EFDD, ο κύριος Μπιτζότο. Η κυρία Μπιτζότο. Στη δεκαετία του 50 και του 60 η θαλιδομίδη δόθηκε στις γύους στην Ευρώπη ως φάρμακο κατά της ναυτίας. Μετά ανακαλύψαμε τι προκάλεσε στην Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία όπου γεννήθηκαν χιλιάδες παιδιά με μεγάλες δυσπλασίες. Σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν 4.000 άτομα τα οποία ζουν ακόμα ε, στο, που ζουν στο πετσί του τη επιπτώσει αυτού του φαρμάκου. Ποιο στέει, μια μεγάλη γερμανική φαρμακοβιομηχανία που δεν ανέλαβε τι ευθύνε τη, αλλά κυρίω στέει και η γερμανική κυβέρνηση, η οποία έκλεισε, έκρυψε την πραγματικότητα για 50 χρόνια και πλέον. Εμεί θέλουμε οι, ε, οι Γερμανοί που είναι οι αφέντε τη Ευρώπη να μην κρύβουν την αλήθεια. Ποιο κρύβει την αλήθεια. Αυτό που κρύβει την αλήθεια είναι συνένοχο. Και το γερμανικό κράτο είναι συνένοχο. Και τώρα α, η Γερμανία ε, κάνει μια κούλπα μπροστά σε χιλιάδε πολίτε. Σήμερα εδώ σε αυτή την αίθουσα μιλάμε για αυτό το πρόβλημα επιτέλου. Αλλά εγώ. Καθώ και η κυρία Τομάσο, η οποία είναι πρόεδρο του Ιδρύματο στην Ιταλία ε, για τα θύματα αυτά, θέλουμε την αλήθεια. Θέλουμε επίσημη συγνώμη από τη Γερμανία, αλλά θέλουμε και αναγνώριση της ευθύνη της με την κατάλληλη αποζημίωση. Φτάνει πια να μας κρύβετε την αλήθεια. Θέλουμε δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη και για τις μητέρες αυτές που αισθάνθηκαν ένοχες αδίκως επειδή πήραν αυτό το καταραμένο φάρμακο. Η κυρία Ντότς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απόψε θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά η στήριξή μας ε, για τα θύματα της τραγωδίας της ε, Θελιδομίδης ε, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί μετά από πέντε δεκαετίες καθώς εξακολουθεί να διατηρεί η τραγωδία τους την σημασία της. Επρόκειτο για ένα φάρμακο για έγκυες ε, γυναίκες και έχουμε άτομα τα οποία στερήθηκαν την ευκαιρία να ζήσουν, μια, να ζήσουν τη ζωή τους ε, στο έπακρο. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από η το κράτος συνεισφέρει μέσω ενός επιδόματος. Όμως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν ο μόνος ένοχος. Πρέπει επιτέλους η γερμανική κυβέρνηση να αναλάβει τις ηθικές της ευθύνες απέναντι στους επιζώντες της ε, Θελιδομήτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ας σοβαρευτούμε. Το κόστος που υπολογίζεται μεταξύ 18 και 25 εκατομμυρίων δεν είναι πολύ για την Γερμανία, αλλά θα σημαίνει τα πάντα για αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζω η συζήτηση αυτή να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στη γερμανική κυβέρνηση πως το ζήτημα αυτό και οι γενναίοι αυτοί άνθρωποι δεν θα εξαφανιστούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος δεν είναι στην αίθουσα. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τραγεδία την, της επληξε έπληξε πολλά κράτη-μέλη και μετά από μισό αιώνα πολλά από αυτά τα θύματα περιμένουν ακόμα αποζημίωση. Η παραγωγή του φαρμάκου, η Grunenthal, η γερμανική εταιρεία, μόνο το 2012 τελικά αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τα χιλιάδε άτομα θύματα, αλλά δεν του δώσε καμία αποζημίωση. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να δώσουμε στήριξη στα θύματα και στι οικογένειέ του. Να προβλέψουμε ένα κατάλληλο πρωτόκολλο, ούτω ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε που είναι θύματα τη ταλιδομίδη να λάβουν αποζημίωση κατάλληλη, ανεξάρτητα από το κράτο μέλο στο οποίο ζουν. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνουν, τόσο ώστε να ζητήσουν μαζί με τα κράτη, από τα κράτη-μέλη μία λύση για να υπάρξει αποζημίωση προς τα θύματα. Τα θύματα και οι οικογένειές τους έχουν απόλυτη ανάγκη από συγκεκριμένη οικονομική στήριξη. Ευχαριστώ. Μαγκίνες. Πόσο χρόνο μου δίνετε, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό που γίνεται αυτή η συζήτηση και θέλω να το χαιρετήσω και ελπίζω να με ε, στρίξετε. Ο Νίκ Ντόμπρικ, ο κύριος Κρέγ Μιλουέρτ και άλλοι πρέπει να τους χαιρετήσουμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν λόμπι και με πίεσαν ε, εδώ το έκαναν με απόλυτη αξιοπρέπεια, με αποτελεσματικότητα, αλλά δεν θα έπρεπε να χρειαζόταν να το κάνουν. Τουλάχιστον πρέπει να αναγνωρίσουμε τη δουλειά που κάνουν, την επιμονή τους και την απόλυτη υπομονή που είναι αυτών που είναι θύματα και που οι άνθρωποι αυτοί τους εκπροσωπούν για να ακούσουν τη φωνή τους. Ε, το πρετανικό δράμα που λέγεται Midwife, ε, ΜΕΑ δηλαδή, δείχνει ε, ένα επεισόδιο για το πώς έτσι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ ουσιαστικά για το πώς ε, γίνεται όταν γεννιέται ένα παιδί ε, με τέτοιες δυσπρασίες. Ε, διάφορες ε, κυβερνήσεις, διαφόρων χρόνων όπου συνέβη, ε, δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε με τη σημερινή συζήτηση. Έχουμε ένα καλό επίτροπο ευτυχώ και είμαστε εδώ δεσμευμένοι, έχουμε την ηθική ευθύνη και το καθήκον να μην αφήσουμε αυτά τα, αυτό το θέμα να ξεχαστεί. Δεν είναι πολλά, πολλά τα λεφτά αυτά η αρχή ότι πρέπει να φροντίσουμε τα θύματα υπάρχει, την έχουμε αναγνωρίσει. Α μην παρετηθούμε μετά από αυτή τη συζήτηση, α προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε με, προς αυτή την προσπάθεια για να τελεσφορήσει αυτή η εκστρατεία και να δοθεί χρηματική αποζημίωση στα θύματα. Ευχαριστώ, ο κύριος Τζοντήλε, η κυρία Τζοντήλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα θύματα της Ταλιδομίδης και η ιστορία τους βαραίνει τις συνειδήσεις μας σαν, ε, με ένα απίστευτο βάρος, βαραίνει τους πρωταγωνιστές, τους θεσμούς και κυρίως όποιος έχει την ευθύνη για να αποζημιώσει ηθικά και οικονομικά τα θύματα αυτά. Ε, στην Ιταλία έχουμε 400 άτομα θύματα. Ε, μερικές χιλιάδες ε, ε θύματα που έχουν πληγεί από αυτές τις, αυτούς τους ακροτηριασμούς που τους καθυλώνουν στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν να ζήσουν μια πλήρη και αξιοπρεπή ζωή. Αυτό το θέμα α, χρήζει της προσοχής μας. Και χαίρομαι τώρα που εδώ στο Κοινοβούλιο συζητάμε τέτοια θέματα που είναι θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Το Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λάβουν μια απόφαση. Να ζητήσουμε συγκεκριμένη δράση από τους πρωταγωνιστές αυτού του δραματικού επεισοδίου. Πέτερλε. Πέτερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συνέβη μια τραγωδία και μια αδικία βεβαίως από την οποία προκύπτουν κάποιες ηθικές υποχρεώσεις. Η αξιοπρέπεια λοιπόν των θυμάτων ε, απαιτεί να αποζημιωθούν για να μπορούν να έχουν μια ποιότητα ζωής ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα βρίσκονται όποιος ε, ήταν θύμα της θαλιδομίδης ε, πρέπει να έχει μία ίση ή ανάλογη τέλος πάντων αποζημίωση από την Κομισιόν λοιπόν που μίλησε με τέτοια ευαισθησία αναμένω και τα ανάλογα μέτρα και να εγγυηθεί ότι θα λάβουν βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα ζουν. Μάθαμε λοιπόν ήδη πάρα πολλά από αυτή την τραγωδία, αλλά λυπούμε για το ότι δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί όλα τα θύματα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ πέρα πως πρέπει να είμαστε συνεπείς. Γνωρίζω τι γινόταν στο παρελθόν. Μιλούσαμε για υγεία, για επιστήμη κτλ. Και μετά τα είδαμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά μπορεί και άλλες ουσίες μετά που θεωρούνται ασφαλείς να αποδειχτούν ε, επικίνδυνες. Ευχαριστώ. Τζοφόλη, στην Ευρώπη οι δραματικές συνέπειες ε, μετά από πάνω από 50 χρόνια από τη χορήγηση σε εγγύους αυτού του φαρμάκου με βάση τη θαλιδομίδη συνεχίζουν να αποτελούν ένα πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους που επέζησαν αλλά η υγεία τους ε, και λόγω της ε, γύρανσης είναι τέτοια που απαιτεί μόνιμη ε, βοήθεια η κατάστασή τους. Με βάση τις πρόσφατες μελέτες που έχουμε, μας έχουν βοηθήσει για να καταλάβουμε τις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων αυτών, μας δείχνουν πόσο αυξημένες είναι οι ανάγκες τους. Πρέπει να δούμε τις αρμοδιότητες που έχουν τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν. Η Κομισιόν πιστεύω και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν θα πρέπει να παρέμβει και να ζητήσει στεναρά μια ισότιμη μεταχείριση όλων, και το υπογραμμίζω, όλων των θυμάτων. Να ξεπεράσουμε τις άδικες διακρίσεις, όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών, αλλά και στο εσωτερικό των ενός ανάλογα με την χρονιά γέννηση. Από το σκάνδαλο τη Θαλιδομίδη, δημιουργήθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των φαρμάκων, για να αποφύγουμε την επανάληψη παρόμοιων δραμάτων. Ακόμα και γι' αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε μόνους αυτούς τους ε, πολίτες μας και τις οικογένειές τους. Σόιντροβα, κυρία Σόιντροβα παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, Ευχαριστώ για την ε, απάντησή σας. Ε, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε το παρελθόν και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν τα σφάλματα. Πρέπει να αποζημιωθούν τα θύματα, ακόμα και αν αυτό βέβαια δεν τους δίνει πίσω την υγεία τους. Είναι όμως κάτι που τους οφείλει το κράτος, η χώρα τους. Τα φάρμακα, η περίθαλψη είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να φεθούν στην ελευθερία της αγοράς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές. Στη Τσεχία το Υπουργείο Υγείας μας ενημέρωσε ότι δεν έχουμε εμεί τέτοιες περιπτώσεις θαλιδομίδης που να έχουν προκαλέσει προβλήματα στην υγεία. Δεν έχουμε τέτοια θύματα. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η Τσεχοσλοβακία δεν χρησιμοποιούσε το φάρμακο αυτό και γι' αυτό δεν έχουμε τέτοια θύματα. Όμως υποστηρίζω τους συναδέρφους μου, τους Ισπανούς, τους Άγγλους, τους Γερμανούς, οι οποίοι μίλησαν υπέρ αποζημίωσης των θυμάτων αυτών. Και πρέπει να πάρουμε και κάποια μαθήματα για το μέλλον. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί κάθε φορά που παράγονται νέα φάρμακα. Η υγεία πρέπει να είναι προτεραιότητα και όχι το κέρδος των φαρμακευτικών εταιριών πεπισμένο ότι έχει καλές πρακτικές η Τσεχία γιατί η πρόληψη είναι πάρα πολύ αυστηρή όταν φέρνουμε στο εμπόριο νέα φάρμακα. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Στήλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τους επιζήσαντες από τη θελειδομή ήδη στην ε, περιφέρειά μου είναι οι ανάγκες που έχουν για φροντίδα που είναι όλο και περισσότερα. Συγκεκριμένα, ένα θύμα, μια γυναίκα μου είπε ότι οι επιλογές στη ζωή της είναι πολύ περιορισμένες. Επιλογές που για άλλους, για όλους εμάς είναι δεδομένες. Δεν μπορεί εύκολα είτε να μπει στο μπάνιο είτε να αλλάξει το παιδί της. Είναι πράγματα τα οποία η γερμανική κυβέρνηση τα γνωρίζει και έχει βοηθήσει 6.000 θύματα και τα βοήθησε να μπουν σε μια νέα περίοδο στη ζωή τους με περισσότερη ποιότητα και να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Σήμερα ζητάμε από τη γερμανική κυβέρνηση να, αφήσουν, να βοηθήσει και τους υπόλοιπους επιζήσαντες ολόκληρη την Ευρώπη. Και χαίρομαι που το θέμα αυτό μας ενώνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώνει όλες τις πλευρές. Και σωστά, όλοι πρέπει να προχωρήσουμε σε εκστρατεία για αυτό το ζήτημα. Και χαίρομαι που βρισκόμαστε στην αρχή μιας εκστρατείας η οποία δεν κυκλοφορεί μόνο στα γραφεία και στους διαδρόμους αλλά και στο σώμα αυτό εδώ στην Ολομέλεια εκεί όπου ανήκει δηλαδή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Καρδίνη, για ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κινήσω όχι με τα δεδομένα τα οποία τα ακούσαμε, τα θυμόμαστε αλλά με τα λόγια του Προέδρου της Οργάνωσης ε, των Θυμάτων της Θαλιδομίδης, που χάρη στην δράση, ε, λέει, ημών των ε, θυμάτων, επινοήθηκε στην Ευρώπη φαρμακοεπαγρύπνηση και υπάρχουν αυστηρά τεστ πριν τεθεί στο εμπόριο ένα φάρμακο. Πέρυσι ήταν η 50η επέτειος του πρώτου νόμου για την φάρμακοεπαγρύπνηση. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί έχουμε να κάνουμε μια πραγματική τραγωδία που κρατάει εδώ και 50 χρόνια ε, με ψέματα, καθυστερήσεις που πλήττουν ε, εκατοντάδες ή και χιλιάδες άτομα και της οικογένειάς τους. Ο Ζιλ Ντελές, ε, Γάλλος φιλόσοφος, έλεγε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα θύματα, αλλά είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στα θύματα. Και απέναντι στα θύματα δεν αρκούν οι δικαιολογίες πρέπει να πληρώσουμε και να ε, αποζημιώσουμε. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε την καταστροφή, αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε μία αποζημίωση, ώστε να τους ε, επιτρέψουμε να αντιμετωπίσουμε με ηρεμία την, ε, τις καθημερινές ανάγκες που λόγω της, των γυρατιών γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Δεν θα πρέπει αυτή η συζήτηση να παραμείνει μόνο στα λόγια. Ζητάω από εσά, Επίτροπε, εξ ονόματος όλων ημών, να μπείτε στο πετσί του διαμεσολαβητή, το ώστε να βρείτε ε, μια λύση ε, ανάμεσα στην γερμανική εταιρεία, το γερμανικό κράτος ε, και τα θύματα, ούτως ώστε όλοι οι πληττόμενοι να βρουν δικαιοσύνη. Η κυρία Σταράς Φαραγκούτα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρασαν πάνω από 50 χρόνια ήδη από το ολοκαύτωμα της Ελίδου Ντροπή το φάρμακο αυτό που πουλιόταν σαν κάτι εντελώς αυλαβές, όπως η ζάχαρη και οδήγησε σε χιλιάδες ανθρώπους με δυσπλασίες. Στη Γαλλία με τον Φράγκο το κρύψαμε. Η δημοκρατία δεν έδωσε απάντηση. Στη συνέχεια όμως είπαμε ότι πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα. Τα εργαστήρια, το γερμανικό για παράδειγμα, αγνόησε και έβαλε τα οικονομικά συμφέροντα πάνω από την ανθρώπινη εξωπρέπεια και την υγεία. Αυτή είναι μια ευθύνη που κάποιο πρέπει να αναλάβει. Γι' αυτό και ζητάμε τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ευθύνη τη φαρμακευτική εταιρεία η οποία έφερε στο εμπόριο το φάρμακο αυτό, αλλά και της γερμανικής κυβέρνησης που επίσης επέτρεψε να κυκλοφορήσει και στο εξωτερικό εκτός Γερμανίας. Και υπάρχει και ευθύνη από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών που επέτρεψαν να κυκλοφορήσει στις χώρες τους το φάρμακο αυτό. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες όπου τα θύματα ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί. Σήμερα λοιπόν εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλά μπορούμε να κάνουμε γιατί έχουμε την ευκαιρία να υποστηρίξουμε την ισότητα να δείξουμε όταν ήκουμε σε μια Ευρώπη η οποία δεν ξεχνάει τους αθώους της. Όταν έχουμε αδέρφια πολλά που υποφέρουν από μια δικία, υποφέρουν, πολλοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, ε, πρέπει να τοποθετηθούμε. Το να μένουμε ουδέτεροι σημαίνει ότι διονύζουμε την αδικία. Αντίθετα πρέπει να βοηθήσουμε τα θύματα. Γι' αυτό ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση. Να μην μείνουμε στα λόγια, αλλά να βοηθήσουμε τα θύματα. Ευχαριστώ. Περνάμε το στο Κατσιάι. Πώς Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη συγκίνηση όλη αυτή την ε, συζήτηση και ευχαριστώ τους συντάκτες που έθεσαν αυτό το θέμα στην Ολομέλεια. Ακούσαμε τρομακτικές αλήθειες, όπου 900 θύματα δεν έχουν αποζημιωθεί. Ε, ακούσαμε ότι κάποιες κυβερνήσεις τους έστρεψαν την πλάτη. Ο Επίτροπος είπε ότι συνάντησε κάποια θύματα και είπε επίσης ότι το πρόβλημα της ε, αποζημίωσης δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστό. Αλλά εδώ εκπροσωπούμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που μας εξέλεξαν σε ελεύθερες εκλογές. Και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να τους δώσουμε απάντηση. Να πιέσουμε τις διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να, να ασχοληθούν με το πρόβλημα αυτό. Επίτροπε, να μην σταματήσουμε σε μια συζήτηση με τα θύματα. Ζητάω από την Κομισιόν να πιέσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την φαρμακευτική αυτή εταιρεία, ούτω ώστε να αποζημιωθούν τα θύματα για να μπορέσουν να ζήσουν με κάθε αξιοπρέπεια. Αγιλέρα Γαρτία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ενώνω τη φωνή μου με τους μαθήτων συναδέλφων που μίλησαν για αυτή την μεγάλη κυρία θύμα της Θαλιδομίδης. Ε, θέλω να μιλήσω για τα θύματα της ε, στην Ισπανία, που δεν έλαβαν καμία αποζημίωση. Έγιναν δύο φορές θύματα. Ε, για αυτά τα θύματα και για την ε, οργάνωσή τους στην Αβίτε, που τα υπερασπίζεται, υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους, και δεν μας κάνει να μην ξεχνάμε αυτό το δράμα. Ε, ακούμε σήμερα στην Ολομέλεια τον κύριο Στέφαν Γκονσάλες και ακούσαμε ότι ε, το Λαϊκό Κόμμα δεν βοήθησε ε, τα θύματα. Ε, οι σοσιαλιστές κάτι κάνανε, όχι αρκετά, αλλά κάτι κάνανε. Αλλά το Λαϊκό Κόμμα δεν έκανε τίποτα. Εδώ και 50 χρόνια και παραπάνω ε, υπάρχει μια τεράστια διακριτική μεταχείριση μεταξύ των θυμάτων της θελιδομίδης στην Ευρώπη και απαιτείται μια ευρωπαϊκή απάντηση. Αλλιώς αυτά τα, τα άτομα θα γίνουν δύο φορές θύματα και αυτό είναι άδικο. Κάντε ό,τι μπορείτε, ε, κύριε Επίτροπε, με ευαισθησία απέναντι στα θύματα. Ειδικά τους Ισπανούς που είναι θύματα, που γεννήθηκαν ανάπηρα, όχι γιατί φταίγαν αυτά. Δεν θα πρέπει λοιπόν, επειδή γεννήθηκαν στην Ισπανία, να γίνουν θύματα δύο φορές. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της θαλιδομίδης μας απασχόλησε αναλυτικά στην Επιτροπή Αναφορών εκεί ήρθαν τα θύματα όπου έθεσαν το ζήτημα. ακούσαμε όλες τις απόψεις και είπαμε ότι πρέπει αυτό το θέμα να προχωρήσει και να προχωρήσει στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου όπως και κάνουμε τώρα διότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί κυρίως την ισπανία όλα αυτά τα χρόνια όπου το καθεστώς του φράγκο κυριολεκτικά έκρυψε το ζήτημα αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση. το ίδιο ισχύει και για άλλα θύματα σε άλλες περιοχές όπως είναι στο βέλγιο στη γερμανία και σε άλλα κράτη. το ερώτημα είναι τι κάνουμε. θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει αποζημίωση των θυμάτων. την αποζημίωση πρέπει να καταβάλει η γερμανική φαρμακευτική εταιρεία όπως επίσης και το γερμανικό κράτος. έχει τεράστιες ευθύνες που δεν έλεγξε το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν που οδήγησε σε παρενέργειες. ευθύνες έχουν και κυβερνήσεις συγκεκριμένων κρατών που κράτησαν το ζήτημα αυτό σε σχέση με την διακίνηση των προϊόντων του φαρμάκου αυτού. επομένως το θέμα είναι επίκαιρο και πρέπει κύριε επίτροπε να έχουμε μια απάντηση μια προσπάθεια και από την κομισιόν παρότι όπως λέτε δεν υπάρχει αρμοδιότητα της επιτροπής στο ζήτημα αυτό. Ο Επίτροπος έχει το λόγο, ο κύριος Ανδρουκάητης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βεβαίως και συμφωνώ απολύτως με όλους σας. Όμως ας ενωθούμε, ας κάνουμε τα πράγματα μαζί. Γιατί εγώ ασχολήθηκα με αυτά τα θέματα, με πυγμή. Έθεσα το θέμα στην φαρμακοβιομηχανία Βεβαίω, δεν είναι αλήθεια να πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα απολύτω. Όχι, κάποια πράγματα έγιναν, αλλά ήταν τα ελάχιστα. Γιατί προκύπτουν και νέα προβλήματα. Πρέπει να δούμε πώς θα στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα. Τι λύση θα βρούμε σήμερα. Θέλω να ακούσω τις ιδέες σας. Πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα αναλύουμε την νομική κατάσταση, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Δεν αρκεί να πει Επιτροπή, λέτε κύριε Επίτροπε κάντε, εντάξει εγώ θέλω να κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Αλλά είναι τόσο δύσκολο. Είμαι γιατρός. Και το καταλαβαίνω. Ίσως μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητήσουμε ξανά με τις εθνικές κυβερνήσεις. Ορίστε, το Συμβούλιο δεν είναι εδώ παρόν. Εσείς μπορείτε να επηρεάσετε, οπότε σας ζητάω και σας να πιέσετε τις κυβερνήσεις σας. Ίσως έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ θα το κάνω. Είναι και υποχρέωσή μου και θα το κάνω. Αλλά χρειάζομαι και από εσά βοήθεια. Θέλω κοινή δράση για το πώς θα προχωρήσουμε, για το πώς ενωμένοι θα προχωρήσουμε. Πριν από δύο εβδομάδες συζήτησα με την φαρμακοβιομηχανία και πάλι και τους ρώτησα είσαστε έτοιμοι να καταλάβετε ότι είναι θέμα εμπιστοσύνη, ότι είναι και θέμα ηθικής ευθύνη. Πώς θα έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος στη φαρμακοβιομηχανία. Λοιπόν, ναι, εγώ είμαι έτοιμος. Στείλτε μου τις απόψεις, κάποιοι αναφερθήκατε στην οδηγία δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με την οδηγία. Φυσικά και πρέπει να ψάξουμε δυνατότητες, μήπως μπορούμε να εισάγουμε νέους κανόνες. Ναι. Δεν αρκεί να κάνουμε δηλώσεις, δεν φτάνει. Δεν φτάνουν τα λόγια, αποτελέσματα χρειάζονται. Και φυσικά και είμαι έτοιμος και είμαι ανοιχτό και θα συνεχίσω να παρακολουθώ το ζήτημα και να ψάχνω να βρω δυνατότητες για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες λύσεις που θα βοηθήσουν τους επιζώντες, τα θύματα. Αλλά όπως είπατε, δεν αφορά μόνο τη γερμανική κυβέρνηση και την ισπανική. Ξέρω ότι η ισπανική κυβέρνηση δεν έκανε αρκετά από τη έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, αλλά μαζί πρέπει να συζητήσουμε. Ιταλία, Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία Γερμανία και ο κλάδος βέβαια, η φαρμακοβιομηχανία για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε πρακτικές λύσεις. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, αλλά ζητάω και από εσά να δραστηριοποιηθείτε, να πιέσετε τις κυβερνήσεις σας, να θέσετε το θέμα και στα εθνικά κοινοβούλια καλέστε και επιτροπές, καλέστε επιτροπές σε εθνικό επίπεδο που είναι αρμόδιες για τέτοια ζητήματα. Δεν αρκεί το blaming and shaming να δείχνουμε με το δάχτυλο δηλαδή το ποιος φταίει. Όλοι μαζί πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τελείωσε η συζήτηση.